Όλες οι ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών που στρέφονται προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώνονται σε ένα κοινό παρονομαστή στον οποίο συγκλίνουν. Είναι το να δούμε τι γίνεται με την κατάσταση των Ρώμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση με αυτό υπάρχει και η δυσφορία η οποία πολλές φορές ε, ε, εκφράζεται όσον αφορά την χρήση κονδυλίων και την χρήση των ε, κονδυλίων για την κοινωνική ένταξη. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι η δράση των ΜΚΟ και αυτά πρέπει να τα δούμε. Είναι σημαντικό να επιστήσουμε την προσοχή ότι πώς ο τρόπος με τον οποίο επιλύονται τα προβλήματα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ας είμαστε ειλικρινείς. Μετά από πολλά χρόνια γενικόλογων και αφηρημένων τοποθετήσεων και μεγαλόστομων διακηρύξεων υπάρχει ανάγκη να γίνουν χειροπιαστά βήματα και δράσεις. Είμαι ανυποχώρητη υπέρ δράσεων και μέτρων για τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων που έχουν συσσωρευτεί αυτά τα αιτήματα εδώ και χρόνια ε, ακούμε τι γίνεται σε σχέση με την αρνητική μεταχείριση των Ρώμα και την ανάγκη να βρεθούν λύσεις στα προβλήματά τους. Μετά από πολλές ε, συζητήσεις δεν είμαστε σε θέση συγκεκριμένα μέσα και συγκεκριμένες λύσεις να εγκριθούν και να υιοθετηθούν. Και είμαι πεισμένη ότι επειδή ε, επικεντρωνόμαστε στον τεχνικό όρο διακριτική μεταχείριση Όλα τα άλλα δεν μπορούμε να τα δούμε και πρέπει εδώ λοιπόν να επικεντρωθούμε στο τι πρέπει να γίνει. Πραγματικά σε σχέση με τα προβλήματα των Ρωμά, θέλουμε να τα λύσουμε, πρέπει να είμαστε υπέρ του, τον, ε, του σεβασμού των ε, διεθνών συμφωνιών και συνθήκων. Για παράδειγμα, τη χάρτα των δικαιωμάτων των παιδιών έχουμε εδώ πολλές φορές παραβίαση των αρχών αυτών των ε, συμφωνιών και συνθήκων. Θα πω τι γίνεται σε σχέση με τη δική μου χώρα, σε σχέση με τα θέματα παιδείας και υγειονομικής περίθαλψης το κράτος παρέχει αυτές τις υπηρεσίες, αλλά και σε αυτές τις πολιτικές τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών δεν γίνονται σεβαστά. Επίσης θα πρέπει, αν θέλουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων, των Ρωμά, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα αίτια τα οποία οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση. Σας ευχαριστούμε. Στη συνέχεια η κυρία Φλότρ, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η Υπηρεσία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λέγουν ότι οι Ρώμα συλλέγουν και υφίστανται όλες τις μορφές διακρίσεων και τους περιορισμούς στην εκπαίδευση και στην υγεία, στη φροντίδα στην υγεία. Ε, γενικά το 2000 ο ένας στους τέσσερις είχε υποστεί επιθέσεις, παρενοχλήσεις σοβαρές και ο ένας στους τρεις είχε συλληφθεί από την αστυνομία τουλάχιστον τέσσερις φορές τον προηγούμενο χρόνο. Η διαδικασία περιθωριοποίησης τους τροφοδοτείται συνεχώς από την έλλειψη ε, γνώσεων σχετικά με τα δικαιώματά τους. Μιλάμε για 10 εκατομμύρια κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα βάλει την υπογραφή της, θα επικυρώσει επιτέλους και τη Διεθνή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις υπόλοιπες χώρες. Χρειάστηκε να υπάρξουν οι ρατσιστικές κινητοποιήσεις του 2007 στην Ιταλία για να καταλήξουμε επιτέλους την οργάνωση της πρώτης συνάντησης κορυφής του Σεπτεμβρίου 2008. Η έκκληση για μια στρατηγική πλαίσιο για την ενσωμάτωση των Ρώμα δεν έχει υλοποιηθεί. Τα κράτη-μέλη σαν τη Γαλλία ε, που ε, έχουν θέσει σε ισχύ μεταβατικά μέτρα για τους Ρωμάνους και τους ε, Ρωμάνους. Τα μέτρα αυτά φύγουν κυρίως τους Ρώμα και θα πρέπει να αναιρεθούν το ταχύτερο δυνατόν. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει επίσης να σταματήσουν τη σύναψη συμφωνιών επαναπροώθησης με το κοσυφοπέδιο γιατί οδηγεί τους ανθρώπους αυτούς να εγκαθίστανται υποχρεωτικά στα βόρεια της Μητρόβιτσα σε περιοχές μολυσμένες από επικίνδυνα χημικά. Να υπενθυμίσω το ψήφισμα της 11ης Μαΐου του 2009 για την κοινωνική κατάσταση των Ρώμα. Φέτος καταπολεμάμε την φτώχεια. Είναι η χρονιά για την καταπολέμηση της φτώχειας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε με τα διαθέσιμα μέσα όπως και τα διαφθρωτικά μέσα για να διορθώσουμε την κατάσταση. Σας ευχαριστούμε εξ ονόματος του Συμβουλίου. Ο κύριος Γιαννίδο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω στις ερωτήσεις που τέθηκαν από την κυρία Φλασίκοβα και από την κυρία Φλότρο σε σχέση με ένα θέμα άμεσα ε, αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και αφορά όλους μας άμεσα και που έχει επιπτώσεις σε ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού γιατί όπως γνωρίζουμε η Τσιγκάνη είναι η πρώτη μειονότητα αριθμητικά που ζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι ακριβώς στο ίδιο επίπεδο διαβίωσης με το μέσο όρο διαβίωση, επίπεδο διαβίωσης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα για τις ερωτήσεις που έγιναν Υπάρχει η πρώτη που κάνει λόγο για την εφαρμογή της χρήσης των διαθωτικών ταμείων σε σχέση ακριβώς με τους τσιγκάνους. Και πρέπει σχετικά με αυτό να σας πω ότι τα συμπεράσματα που η Ισπανική Προεδρία πρόκειται να υιοθετήσει στο Συμβούλιο συμπεριλαμβάνουν αυτές τις δέκα βασικές αρχές μεταξύ των οποίων είναι η αναθεώρηση, η κωδικοποίηση των υφισταμένων λειτουργικών προγραμμάτων των ε, διαθωτικών ταμείων καθώς επίσης και οι μελλοντικοί κανονισμοί από το 2014 και εφ' εξής. Και υπάρχει, εμένουμε να γίνεται πλήρης ε, χρήση των διαθωτικών κονδυλίων για την ένταξη των συγκάνων των Ρωμά. Συγκεκριμένα προτείνουμε να λειτουργήσουν, να δρομολογηθούν δράσεις ε, στις αστικές και ε, υπαίθριες περιοχές σε σχέση με το άρθρο 7 του ΦΕΝΤΕΡ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Και έτσι οι κοινότητες των Ρώμα να έχουν καλύτερη δυνατότητα στέγασης και κοινωνικής διαβίωσης. Και όσον αφορά τις τοπικές αρχές. Εμείς θεωρούμε ότι για να μπορέσουν τα διαθωτικά ταμεία να είναι προσπελάσιμα, προσβάσιμα στους Ρωμά, στους Τσιγκάνους, πρέπει να αναπτυχθούν δράσεις των τοπικών αρχών, καθώς επίσης και των ίδιων των οργανώσεων των Τσιγκάνων, καθώς επίσης και την εμπλοκή των Τσιγκάνων σε όλη τη διαδικασία, από τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των δράσεων των κονδυλίων των Ευρωπαϊκών Διαθωτικών Ταμείων. Επίσης ε, το ε, Συμβούλιο θα ήθελε Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεπικουρεί τα κράτη-μέλη και τις τοπικές αρχές στην υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων και να υπάρξει η διευκόλυνση οριζόντιου συντονισμού και κάθε του επίσης συντονισμού μεταξύ του τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και ευρωπαϊκού επίπεδου. Μια τρίτη ερώτηση αφορά αν η Προεδρία έχει μια στρατηγική πρόταση ή ένα στρατηγικό σχέδιο σε σχέση με την πολιτική για τους τσιγκάνους. Θα ήθελα να σας πω ότι στο πρόγραμμα της ε, τριπλής ε, προεδρίας των, των ε,

τριών προεδριών γίνεται λόγος για την κοινωνική ένταξη ε, των συγκάνων. Είναι μια έκφραση που έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και ομόφωνα και γι' αυτό ανταποκρίνεται ακριβώς στη στρατηγική για το επόμενο 1,5 έτος ε, για την ε, διάρκεια δηλαδή του προγράμματος της τριπλής προεδρίας αλληλοδιάδοχων τριών προεδριών. Υπάρχουν λοιπόν βραχυπρόθεσμα μέτρα, βραχυπρόθεσμα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στα μέτρα εκείνα στα οποία προαναφέρθηκα μόλις το πριν και να υπάρξει η έγκριση ενός προγράμματος εργασίας ώστε άμεσα να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως π.χ. των μαθητών που πάνε σε ειδικά σχολεία, σε κάποιες περιπτώσεις και μάλιστα αποκλειστικά σχολεία τσιγκάνων. Και πρέπει να αποφύγουμε τον ε, διαχωρισμό, τον αποκλεισμό και επίσης να δούμε και το θέμα της στέγασης και των υγειονομικών ε, ε, υπηρεσιών που θα παρέχονται στους τσιγκάνους μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και να υπάρξει και μια οριζόντια επικέντρωση mainstreaming όλων των πολιτικών δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να συμπεριλαμβάνουν τα θέματα των τσιγκάνων όπου χρειάζεται και η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού και η αντιμετώπιση της αρνητική διακριτικής μεταχείρισης και όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση καθώς επίσης και την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες ευρύτερα. Και τέλος να προσθέσω ότι όσον αφορά τα θέματα μη αρνητική ε, μεταχείριση. Γνωρίζετε ότι η Ισπανική Προεδρία καταβάλει προσπάθειε να προαγάγει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου τη και στην τριπλή μορφή των ε, εναλλασσομένων Προεδριών την έγκριση. Θέλει να πετύχει μια οδηγία που εδώ και χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε καταφέρει να εγκρίνουμε, που είναι η ολοκληρωμένη οδηγία για την καταπολέμηση τη αρνητική διακριτική μεταχείριση και τη ε, μη ίση αντιμετώπιση. Ιδιαίτερη σημασία για εκείνες τις μειονότητες ε, που υφίστανται αρνητική μεταχείριση και ιδιαίτερα για τους Ρωμά, του Τσιγκάνου. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Λόπες Γκαρίδο. Γκαρίδο. Εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επίτροπος Ρέντινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σβόβοντα και τους συναδέλφους τους επειδή κατέθεσαν αυτή την προφορική ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τους Ρωμά. Δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκφράσει τη δέσμευσή της για να διασφαλίσει ότι ε, θα τηρούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα αφενός και ε, θα γίνουν προσπάθειες για την οικονομικη ένταξη τους ε, στην κοινωνία μας αφετέρου. Μόλις ακούσαμε το Συμβούλιο, το οποίο δεσμεύτηκε πραγματικά ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προχωρήσουν το θέμα αυτό τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και να το συμπεριλάβουν στις πολιτικές τους. Ξέρετε ότι η συζήτηση αυτή γίνεται λίγες εβδομάδες ε, πριν από τη δεύτερη διάσκεψη των Ρωμά που θα γίνει στην Κόρδοβα. Ε, θα είναι η Ισπανική Προεδρία στις 9 ε, Απριλίου και χαιρετίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την πρωτοβουλία. Θεωρούμε ότι θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να δούμε πώς έχουν προχωρήσει οι εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. να δούμε τι έγινε από το 2008 και θα μας βοηθήσει και να συνεισφέρουμε σε, ένα, σε μια πολύ καλή προοπτική για το μέλλον. Πριν από δύο χρόνια είχαμε την πρώτη διάσκεψη. Πού φτάσαμε στο μεταξύ ο καθένα μπορεί να βλέπει το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο. Σαφώ έχουν γίνει πολύ ουσιαστικέ βελτιώσει, ωστόσο υπάρχουν και πολύ ουσιαστικά κενά. Και αυτή τη στιγμή επισημαίνεται ο κεντρικός ρόλος των ε, μέσων και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σημασία του να ενισχύσουμε τη συνεργασία, τη συνεργασία μεταξύ όλων των βασικών ε, συμμετεχόντων, ε, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, διεθνών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να εφαρμόσει μια οδηγία η οποία απαγορεύει τη διάκριση για λόγους φύλου και εθνικής ε, καταγωγής και η διάκριση κατά τον Ρωμά καλύπτεται από αυτή την οδηγία. Υπάρχει και ποινικό δίκαιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η απόφαση πλαίσιο για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, που θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε τον ρατσισμό από τον οποίο πλήττονται οι Ρωμά. Όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θέσουν, ε, να δημιουργήσουν ποινικέ κυρώσεις ε, για αδικήματα ε, ξενοφοβίας και ρατσισμού βάσει της απόφασης πλαίσιο και όπως σας ανακοίνωσα ήδη είμαι διατεθειμένη να παρακολουθήσω την εφαρμογή αυτής της απόφασης πλαίσιο όσο το δυνατόν πιο στενά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνειδητοποιεί βέβαια πλήρως ότι αυτό δεν επαρκεί και θα πρέπει να υπάρξουν και συμπληρωματικά μέτρα και να υπάρχει δυνατότητα πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για τα θέματα αυτά. Και προς αυτό το σκοπό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τα θέματα των Ρωμά και υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την ποικιλο... Ε, μορφία και τις συγκεκριμένες πρακτικές ε, για τους νομικούς. Αυτή τη στιγμή τα διορθωτικά ταμεία και τα ταμεία ανάπτυξης, ε, όπως επίσης και τα μέσα προενταξιακής βοήθειας, αποτελούν πολύ σημαντικού μοχλούς για τι αλλαγέ, διότι επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν φιλόδοξα προγράμματα, τα οποία στοχεύουν στου Ρωμά συγκεκριμένα. Και είναι δεδομένο ότι τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να είναι πολύ ρεαλιστικά και να βασίζονται σε απτά στοιχεία. Σαφώ θα πρέπει να προσεγγίζουν το, οι συνθήκε διαβίωσης των Ρωμά και να βλέπουν το θέμα με όλε τι πολύπλοκε πτυχέ του. Διότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε απλά, να χρησιμοποιούμε απλά λόγια για να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο ζήτημα χρειαζόμαστε συγκεκριμένες πράξεις. Γι' αυτό ακριβώ και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πλήρω τα ταμεία αυτά για να υποστηρίξουμε την ενσωμάτωση των Ρωμά. Έχουν ξεκινήσει και μια σειρά από υψηλού επίπεδου επισκέψεις διμερώς ε, στα κράτη-μέλη και θα συναντήσουμε και πληθυσμούς Ρωμά και θα προσπαθήσουμε να έχουμε συγκεκριμένους συμπεφωνημένους στόχους. Η πρώτη επίσκεψη έγινε τον Οκτώβριο του 2009 στην Ουγγαρία με πλήρη συνεργασία της κυβέρνησης και θα οργανωθούν και άλλες στο μέλλον. Ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα τη δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρήση των διαφορετικών ταμείων για την καταπολέμηση των αποκλεισμού των Ρωμά είναι οι τροπολογίε που ε, προτάθηκαν για το άρθρο 7, παράγραφος 2, του, Ευρωπαϊκού Ταμείου, του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και η αθρώα πλειοψηφία που ψήφισε εδώ στην Ολομέλεια την έκθεση του συναδέλφου σας, του κυρίου Φαν Λίστεροι, στις αρχές του περασμένου μηνός, δίνει τη δυνατότητα ε, για νέα χρηματοδότηση και νέα πολιτική για τη στέγαση ε, προς των περιθωριοποιημένων κοινωνιών. Και μπορούμε λοιπόν να στοχεύσουμε συγκεκριμένα στους Ρωμά, αλλά όχι μόνον σε αυτούς. Τέλος, χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν και πιλωτικά προγράμματα για την ε, ενσωμάτωση των Ρωμά. Υπάρχει ένας προϋπολογισμός 5 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος θα κατανεμηθεί σε δύο έτη. Ε, μας αφορά η παιδεία στη μικρή πελική ηλικία και η ευαισθητοποίηση του κοινού. Η αξιολόγηση αυτών των πιλωτικών προγραμμάτων θα γίνει από κοινού μεταξύ ε, του UNDP και της Παγκόσμιας Τράπεζας και προσβλέπω σε αυτή την αξιολόγηση γιατί η αξιολόγηση θα μας δώσει τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να γνωρίζουμε τι κάναμε σωστά και πού υπάρχουν οι ελλείψεις ώστε να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά προκειμένου να προχωρήσουμε με πολύ στοχευμένες δράσεις ε, στη συνέχεια. Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τη Μεσομάτωση των Ρωμά ε, ξεκίνησε ως κοινή πρωτοβουλία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Τσεχικής Προεδρίας το 2009 και στόχος είναι να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι σε ευρωπαϊκό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και ενδιαφερόμενοι από την κοινωνία των πολιτών και οι υφιστάμενες πολιτικές να γίνουν όλο και περισσότερο συνεκτικές. Η πλατφόρμα αυτή έχει οδηγήσει στην εκπόνηση των βασικών αρχών για την ενσωμάτωση των Ρωμών, που αποτελεί παράρτημα στα συμπεράσματα της συμπερίληψης των Ρωμά που υιοθετήθηκαν από τα Υπουργικά Συμβούλια τον Ιούνιο πέρσι. Τα συμπεράσματα αυτά καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις 10 βασικές αρχές για τη συμπερίληψη των Ρωμά όταν θα σχεδιάζει και θα εφαρμόζει πολιτικές αναμένεται να υπάρξουν και άλλες συναντήσεις της πλατφόρμας στη διάρκεια της Ισπανικής και της Βελγικής Προεδρίας. Επομένως δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνεται περιστασιακά. Πρόκειται για μια δράση η οποία παρακολουθείται στενά και Χαιρετίζω τη δέσμευση του Στρόικα των Προεδρών για τον στόχο αυτό, κύριε Πρόεδρε, διότι Θεωρώ ότι το ένα χέρι είναι βιτάλο και θα πρέπει να ε, βοηθάμε ο ένα τον άλλον να συνδράμουμε προκειμένου να προχωρήσει το θέμα αυτό. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συνεισφέρει στι δράσει της Τρόικα για να έχει φυσικά και στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη και την κοινωνία των πολιτών. Εν ώψη λοιπόν της διάσκεψης των Ρωμά θα ήθελα να ενημερώσω τη, κύριε Πρόεδρε το Κοινοβούλιο ότι θα δημοσιεύσουμε μια ανακοίνωση για την ένταξη των Ρωμά θα επισημάνουμε τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσει τις, προσκλη... τις προκλήσεις και φυσικά αυτό θα αποτελέσει και τη βάση της συζήτησης στην Κόρδοβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Να περάσουμε τώρα στους ομιλητές εξ ονόματος των ομάδων. Θα ήθελα να τηρήσετε το χρονοδιάγραμμα, διότι στις 6 έχουμε το γύρο των ερωτήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν μας πιέζει λίγο χρόνος. Εξ του ΕΛΚ, για δύο λεπτά, η κυρία Ζάροκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η καταπολέμηση της διάκρισης απαιτεί πιο αποτελεσματικά μέτρα για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρωμά. Τα κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια έχουν ε, δει ότι υπάρχουν πολλά σχέδια και πολλών ε, διεθνών οργανώσεων, αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί αυτά τα σχέδια για πολλούς λόγους και οικονομικούς μεταξύ άλλων. Ε, υπάρχει και το λεγόμενο soft law, το ήπιο δίκαιο, ε, με κοινού δείκτε και με κοινέ προσπάθειες. Ω εισηγητρία εγώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Ρωμά, Γνωρίζω ότι χρειάζεται ε, άμεση δράση ε, και λαμβάνοντα υπόψη και τις διαφορές ανάλογα με τη γεωγραφική περιφέρεια. Πολλές φορές οι Ρωμά κατοικούν σε μέρη που έχουν πολύ μεγάλη φτώχεια και πολύ μεγάλο κοινωνικό αποκλεισμό. Είναι πρόκληση για την Ευρώπη. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν ευκαιρίες ε, για τη μειονότητα αυτή με προγράμματα για την ανάπτυξή τους. Η κουρικότητα και απαιτεί να ασχολούνται οι τοπικοί φορείς με την αξιολόγηση και την εφαρμογή της ε, στρατηγικής αυτής. Και όπως γίνεται και με τη Γεωργία, ε, θα πρέπει να κάνουμε επιτόπου επισκέψεις για να διαπιστώνουμε την κατάσταση των ε, ανθρώπων αυτών, καλές οι στατιστικές, καλά τα τεχνικά στοιχεία, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι να ε, τα προσέξει αυτά η Σύνοδος Κορυφής της Κόρδοβας. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Μωράες, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπαν και προηγούμενοι ομιλητές και οι επιτροπού, το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Εκτός από την ερώτηση που θέσαμε σήμερα για τη δική μου την ομάδα και για όλες τις ομάδες πιστεύω πρέπει να ανανεώσουμε και να θερμάνουμε τη συζήτηση για το ζήτημα των Ρωμά. Εδώ η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει απαράδεκτα επίπεδα προκατάληψης και κάποιες φορές και βίας. Είμαστε στη δεκαετία της κοινωνικής ένταξης στο Ρωμά και της σχετικής πρωτοβουλίας και υπάρχει ένα αυξανόμενο αίσθημα σε αυτό το σώμα ότι χρειάζεται μια εδώ συνολική οργανωμένη προσέγγιση. Έχουμε συζητήσει αυτή τη συνολική και ενιαία προσέγγιση και στο παρελθόν. Και έχουμε δει τι πρέπει να γίνει σε σχέση με τις μικροπιστώσεις, την αντιμετώπιση της βίας, αυτά τα πολύπλοκα ζητήματα. Για όλα αυτά χρειάζεται μια συνολική στρατηγική. Έχουμε όλο ένα και περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία ότι η κατάσταση στην πράξη δεν βελτιώνεται αρκετά. Βλέπουμε να μιλάμε για προκαταλήψεις, για φαινόμενα βίας, για κοινωνικό αποκλεισμό κοινοτήτων σε όλη την Ευρώπη και ε, το, ο Οργανισμός για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα έχει επισημάνει φαινόμενα κατά, διακριτικής μεταχείρισης κατά τον Ρωμά περισσότερο από κάθε άλλη μειονοτική ομάδα η υφιστάμενη κατάκταση και με τις υπάρχουσες οδηγίες του Συμβουλίου και τον σχετικό κανονισμό θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Χρειαζόμαστε συνολική εκστατική. Υπόθηκε και προηγουμένω. και πρέπει το θέμα αυτό να το δούμε ως ένα πολυσύνθετο πρόβλημα. Αλλά απαιτείται δράση και μια ε, ενιαία κίνηση, μια συνολική δράση Πρέπει να αναθερμανθεί όλη η συζήτηση, να ανανεωθεί και να εξέφουμε νέε λύσει. Να υλοποιηθούν οι υπάρχοντε νόμοι. Οι νόμοι που θα πρέπει να, ευ... να ευνοήσουν τι κοινότητε των Ρωμά. Για ένα λεπτό το λόγο έχει τώρα ε, η, κυρία Βέμπερ, εξ ονόματος των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εν ώψη της δεύτερης συνόδου κορυφής για τους Ρωμά, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές ιδέες και ελπίζω αυτές το συντομότερο να ελοπιθούν. Προσωπικά πιστεύω στεναρά ότι χρειαζόμαστε μια ευρεία και συνεκτική στρατηγική για τη συμπερίληψη των Ρωμά Επίσης, πρόγραμμα δράσης χρειαζόμαστε με σαφή benchmark για συγκριτική αξιολόγηση και καλή ε, κατάλληλη πρικοδότηση. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τα κράτη-μέλη της Ένωσης, αλλά και για άλλες χώρες που ζουν κοινότητες Ρωμά, είτε στη διαδικασία διεύρυνσης, είτε στη πολιτική γειτονία είναι χώρες αυτές. Και έτσι θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει τα καλύτερα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για τις πολιτικέ για τους Ρωμά. Δεύτερον, θα πρέπει πιστεύω να... Ε, ε, εφαρμόσουμε ό,τι διδαχτήκαμε και από την ισότητα των φύλων. Το mainstreaming, η συμπερίληψη της πολιτικής για τους Ρωμά σε όλες τις εγκάρσεις πολιτικές. Τρίτον, ε, πραγματογνωμοσύνη. Θα πρέπει να κάνουμε ε, κάποιες θετικές διακρίσεις ε, προσλαμβάνοντας τα τρία θεσμικά όργανα Ρωμά για να γνωρίζουμε καλύτερα την κατάσταση. Γι' αυτό προετοίμασα μια επιστολή προς τον πρόεδρο Φαν Ρόμπα και Μπαρόσο να δώσουν το παράδειγμα οι ίδιοι ε, διορίζοντας υψηλό βαθμούς Ρωμά. Από τους Πρασίνους και την Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία, για 1,5 λεπτό η κυρία Λάμπερτ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρου τη ομάδα μου ήθελα να καλωσορίσω τι εκκλήσει που έγιναν και από του υπόλοιπου συναδέλφου για μια συνολική στρατηγική. Όπω ήδη επισημάνθηκε, βρισκόμαστε στο Ευρωπαϊκό Έτο για την καταπολέμηση τη ένδυα και του κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι δύσκολε οι στιγμέ που ζούμε τη οικονομική ύφεση και γι' αυτό ζητούμε να υπάρχει η λήψη υπόψη των κοινωνικών προποθέσεων για να δοθούν πακέτα ενίσχυση. Αυτοί που είναι περισσότερο αποκλεισμένοι από όλου δεν θα πρέπει να είναι ακόμη περισσότερο μειονεκτούντε. Ενώ τα χάσμα και οι διαφορέ μεταξύ των πολιτών μεγαλώνουν. Έχουμε και τη στρατηγική 20 επί 20 τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει να λάβει επίση υπόψη την ανάγκη να καλυφθούν οι διαφορέ μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Οι αλλαγέ ε, στα περιφερειακά ταμεία και στα, και στα διευθυντικά ταμεία είναι σοβαρέ. Βλέπουμε ότι η συνεργασία των επιμέρους αρχών με το Συμβούλιο είναι σημαντική. Γιατί η στέγαση, οι συγκεκριμένε ανάγκε των πληθυσμών των Ρωμά στι διάφορε επαρχίε και τι διάφορε περιφέρειε είναι σημαντικέ. Η εκπαίδευση, η δράση τη αστυνομία που πρέπει να προστατεύει και όχι μόνο να επιβάλλει ε, κυρώσει ή να καταδιώκει. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Θυμάμαι, θυμόμαστε την ε, σύσταση για την ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας στον Ρωμά. Και αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να ξέρουμε εάν η Επιτροπή και το Συμβούλιο είναι ικανοποιημένοι με το ποσοστό απορροφητικότητας που παρουσιάζεται σε σχέση με τα διευθυντικά ταμεία και τα περιφερειακά ταμεία. Η Επιτροπή μιλάει για δράση κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Ελπίζω ότι κάθε κυβέρνηση, κάθε κράτος μέλους θα δεσμευτεί στα ιδανικά που έχει πρεσβεύσει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ από τους ε, συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Για δύο λεπτά ο κύριος Βαντάλεν παρακαλώ. Πρόεδρε, καλό είναι και χρήσιμο το Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με τη μοίρα των Ρωμά. Στους τελευταίους αιώνες η διάκριση ήταν το, το λιγότερο κακό που του συνέβαινε. Ευρωπαϊκά ταμεία, ευρωπαϊκές οδηγίες, καλό είναι να χρησιμοποιηθούν υπέρ τη ένταξη των Ρωμά και της καταπολέμησης καθυστέρηση. Ελπίζω να υπάρξει και μια καλή στρατηγική έτσι ώστε τα ευρωπαϊκά εκατομμύρια πραγματικά να φτάσουν στους πραγματικούς δικαιούχους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση, στην παιδεία. Ε, θα πρέπει να εξοπλιστούν τα παιδιά αυτά με εφόδια για να σπάσουν το φαύλο κύκλο. Θα ήθελα να προσθέσω δύο στοιχεία, Πρόεδρε, και εγώ σημερινή συζήτηση. Πρώτον, δεν θεωρώ καλό το γεγονός ότι παραμένουν πολλοί Ρωμά ε, στην κατάσταση και στην εικόνα του θύματος. Θα πρέπει και οι ίδιοι να αναβάνουν κάποια δράση για να ε, σπάσουν οι προκαταλήψεις και η αρνητική μεταχείριση στην κοινωνία. Και δεύτερον, τα ευρωπαϊκά χρήματα και η ευρωπαϊκή ε, νομοθεσία για τη συμπερίληψή τους δεν μπορούν να επιβληθούν εκ των άλλων. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν την πρωτοβουλία, γιατί στο κάτω-κάτω εκεί ζουν αυτοί οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια, για να του ενσωματώσουν στις κοινωνίες. Είναι περισσότερο κοινωνική αυτή η πρόκληση και λιγότερο πολιτική ή οικονομική. Τα ευρωπαϊκά ε, χρήματα ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, κύριε Πρόεδρε, όμως ως μία όθηση και μόνο. Ευχαριστώ. Από την ε, Ενωτική Αριστερά τώρα το λόγο έχει η κυρία Κορνέλια Έρνστ για 3,5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Το Δεκέμβριο του 2009 πήγα στην Πρίστινα και στη Μητροβίτσα και είδα τους ανθρώπους πώς ζουν στους μαχαλάδες και ε, στους καταβλισμούς που είναι μολυσμένοι από μόλιβδο. και ε, συγκλονίστηκα ιδιαίτερα από τις συνθήκες που επικρατούν και πώς ζουν τα παιδιά. Και έκανα επαφές εκεί και συνομιλίες και έμαθα ότι αυτό δεν ισχύει μόνο στο Κωσυφοπέδιο αλλά και σε άλλες χώρες και είναι από τους πιο ε, παλιούς πληθυσμούς στην Ευρώπη. Από το εκεί, ε, Σουλά και το κέντρο τεκμηρίωσης Ασκάλης στην Πρίστινα έμαθα ότι έχουμε κουραστεί μας λένε οι άνθρωποι αυτοί από τα λόγια. Έργα χρειαζόμαστε τώρα. Και γι' αυτό έχουν αναποθέσει όλες τις ελπίδες τους στην Κόρδοβα. Όχι μόνο ρυθμίσεις, άμεση δράση χρειάζεται. Τι σημαίνει άμεση δράση. Σημαίνει να μην επαναπευθούμε πίσω από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ίση μεταχείριση ε, χωρίς διάκριση εθνικής προέλευσης και φυλής, ούτε και για την οδηγία της απασχόλησης. Δεν βοηθάει αυτό. Χρειάζεται άμεση δράση, επαναλαμβάνω, για να καταλάβει ο κόσμος να αναγνωρίζει ότι οι οδηγίες αυτές δεν αρκούν για να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι Ρωμά και να προστατεύονται από ταπεινωτική και διακριτική μεταχείριση και ε, να το λύσουμε αυτό το θέμα ε, με τρόπο βιώσιμο. Χρειάζεται μια στρατηγική για τους Ρωμά στην Ευρώπη που να σέτε σε όλους τους τομείς της πολιτικής, να είναι ενσωματωμένοι παντού. Οι περισσότερες κυβερνήσεις μόνο προγράμματα υλοποιούν και σποραδικά μέτρα. Αυτό που χρειάζεται όμως είναι μέσω μακροπρόθεσμη πολιτική οικονομικά μέτρα για την οικονομική ανάπτυξη των κοινοτήτων Ρωμά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια της και τα περιφερειακά και τα διορθωτικά, όχι από το 2013 και μετά. Από τώρα να τα αξιοποιήσουν οι Ρωμά, μικροπιστώσεις που να χορηγούνται ε, χωρίς γραφειοκρατία για την ε, ανακαίνιση των καταβλισμών ε, για θέματα δημόσιας υγείας, παιδείας, εκπαίδευσης, προώθησης αγοράς εργασίας. Και το λέω ειλικρινά, κανένα παιδί δεν θα πρέπει να ε, αποτυγχάνει για λόγους ε, παιδείας ή γλώσσας. Και δεν θέλουμε ειδικά σχολεία για τους Ρωμά, θέλουμε να πηγαίνουν στα ίδια σχολεία με όλους. Και κατά τα άλλα αυτό που μας ενδιαφέρει δεν μόνο τα χρήματα, αλλά η καταπολέμηση του ρατσισμού και του αντιτσιγκανισμού να είναι ποινικά κολάσιμο αδίκημα, να μην είναι παράπτωμα ή πλημέλημα αυτή η συμπεριφορά. Ελπίζω το συντομότερο να ανταποκριθούμε και να δικαιωθούν οι Ρωμά στην Ευρώπη που είναι πάνω από 10 εκατομμύρια. Να αρχίσουμε από τη δικαίωσή τους και θα συνεχίσουμε με την εξίσωσή τους. Γι' αυτό χρειάζεται μια πολύ σημαντική πολιτική απόφαση, ένα μεγάλο ναι ε, για την καταπολέμηση της ε, στρατηγικής της στόχης. Και πραγματικά με πάθος με ενδιαφέρει αυτό το θέμα, όχι μόνο ως βουλευτή, αλλά και ως άνθρωπο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δράσουμε υπέρ των Ρωμά και Σίντι. Ευχαριστώ κύριε Ένστ. Εξ ονόματο της Ομάδα Ελευθερία και Δημοκρατίας. για μισή λεπτό ο κύριο Πάσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η δεύτερη σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωμά θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ανταλλάξουν απόψεις και μέτρα για την ενσωμάτωση των Ρωμά στην κοινωνία. Οι πρόγονοι μας πιστεύουν ότι οι Ρωμά έφτασαν ε, στην Ευρώπη μεταξύ του 5ου και του 1 ου αιώνα και έκτοτε όλοι προσπαθούν να εξεύρουν ένα καλύτερο τρόπο συνύπαρξης μεταξύ Ευρωπαίων και Ρωμά. Μετά από χίλια χρόνια και αναζήτησης φαίνεται ότι δεν έχει ακόμα βρεθεί ένας τρόπος ε, σωστής ε, ένταξή του στην κοινωνία μας. Δεν ξέρω αν ε, το φταίξιμο βαραίνει εμάς ή τους Ρωμά. Από την πείρα όμως που έχω στη χώρα μου, γνωρίζω ότι η προσπάθεια να συνδράμουμε μέσω δωρεών δεν θα βοηθήσει. Στη χώρα μου οι πολίτες φορολογήθηκαν σε πολύ υψηλό επίπεδο και δόθηκαν κονδύλια στους Ρωμά από αυτή τη φορολόγηση για να μπορέσουν να έχουν όλοι ένα σπίτι. Ε, δόθηκε πρόσβαση σε απασχόληση και ε, παιδεία ε, και εξισώθηκαν με όλους τους υπολείπους πολίτες. Λαμβάνουν τα ίδια επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης. Αλλά δείτε τα αποτελέσματα. Οι νέες κατοικίες που τους δόθηκαν καταστράφηκαν γίνονται συνεχώς κλοπές, καταστροφές, ε, σε εξοπλισμό ε, ε, αφήνουν απορρίμματα παντού. Πολλές φορές ε, ιατρικό προσωπικό πηγαίνει σε χωριά Ρωμά και τους ε, διώχνουν ε, και τα παιδιά των Ρωμά φεύγουν από τα σχολεία. Εάν θέλουμε λοιπόν να αλλάξει η κατάσταση θα πρέπει να μάθουμε στα παιδιά των Ρωμά να είναι πολιτισμένα. Ευχαριστώ για δύο λεπτά. Ο κύριος Μπάλτσκο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα μιλήσω ουγγρικά τη μετρική μου γλώσσα και θα χρησιμοποιούσα τον όρο αντί για τον κλασικό όρο Ρωμά, γύφτος στη δική μου γλώσσα. Δεν υπάρχει εδώ κάποια διάθεση όμως να εκφραστώ άσχημα. Η κοινωνική ένταξη των Ρωμά, ε, των Ρωμά ε, είχε να κάνει με την ε, άσκηση διακριτικής μεταχείρισης εναντίον τους, ιδίως στην αγορά εργασίας. Αυτό ήταν κάτι που θέλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουν προσπαθήσει να καταπολεμήσουν αυτή τη διάκριση και να περάσουμε σε άμεση ένταξη το Ρωμά. Στην Ουγγαρία έχουμε πολλούς τέτοιους πληθυσμούς που προσπαθούν να ξεφύγουν από αυτό το φαύλο κύκλο αλλά δεν τα καταφέρνουν ιδίω λόγω της δικής μας οικονομικής πολιτικής στην Ουγγαρία. Οι Ρωμά εκπροσωπούν ένα πολύ υψηλό ποσοστό των ε, όσων ασκούν εγκληματικές δραστηριότητες. Τους έχουμε αποτρέψει όχι μόνο για το καλό της ευρύτερης κοινωνίας, αλλά για να είναι σαφές ότι και οι Αθήγανοι μπορούν να είναι έντιμοι και αυτό να φανεί προς τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν μπορούμε εδώ να μιλάμε για γενετικά ή εθνοτικά χαρακτηριστικά και να μην σκεφτόμαστε αμέσως τη διακριτική μεταχείριση. Και βεβαίως αυτό επιφέρει και κοινωνική μειονεξία. Δεν μπορούμε να στιγματίζουμε διαρκώς αυτές τις κοινότητες με μόνο επιχείρημα τον ρατσισμό, αλλά δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι αυτό είναι και το μόνο πρόβλημα. Πρέπει να αναζητήσουμε διέξοδο. Οι ίδιοι οι Ρωμά χρειάζονται αξιόπιστου ηγέτε, πρόσωπα τα οποία οι ίδιε οι μειονότητε να τα αναγνωρίζουν ω εκπροσώπου του, για να γίνουν δεκτοί στα πλαίσια, στου κόλπου τη ευρύτερη κοινωνία. Χρειάζεται εδώ μια ευρωπαϊκή στρατηγική. Μια στρατηγική που να εντοπίζει όλες τις πτυχέ αυτού του προβλήματο. Ευχαριστώ. Να περάσουμε στου υπόλοιπου ομιλητές. Για δύο λεπτά ο κύριος Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώ την παρέμβασή μου δίνοντας συγχαρητήρια για τη μάχη που δίνεται υπέρ των ε, ε, Ρωμά ε, εξ ονόματος ε, της κοινωνίας των Ρωμά. Να υπενθυμίσω ότι το ΕΛΚ ήταν το πρώτο το οποίο ξεκίνησε μια δράση ε, μέσω της κυρίας Γιαρόκα υπέρ των 10 εκατομμυρίων Ρωμά που διαμένουν στην Ευρώπη. Η κατάσταση των Ρωμά είναι διαφορετική των άλλων μειονοτήτων που διαμένουν στην Ευρώπη, γι' αυτό ακριβώς και θα πρέπει να λεφθούν συγκεκριμένα μέτρα που θα αφορούν αυτούς και μόνον αυτούς. Η δεύτερη σύνοδος κορυφής ε, για τους Ρωμά θα πρέπει να αποτελεί το φόρουμ στο οποίο θα ληφθούν μέτρα που θα βοηθήσουν την κοινότητα αυτή και θα είναι πολύ συγκεκριμένα τόσο χρηματοοικονομικά όσο και νομικά ε, για να βοηθήσουν μία μειονότητα η οποία θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει στο, ε, στο ίδιο της το μέλλον. Δεν θα πρέπει να έχουμε μία πατερναλιστική πολιτική και δεν έχει κανένα το δικαίωμα να κάνει πολιτική διαφήμιση ε, εις βάρος τους. Μόνο μια συντονισμένη πολιτική μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κοινοβουλίου και κρατών μελών θα δώσει θετικά αποτελέσματα υπέρ των Ρωμά. Οι διάφοροι ε, Ευρωπαίοι Επίτροποι θα πρέπει να συντονιστούν ώστε να καθορίσουν και να διευκρινίσουν ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία διακριτική μεταχείριση θα πρέπει το Συμβούλιο μαζί με τα κράτη-μέλη να επιβεβαιώσει ότι θα υπάρχει πλήρη ενσωμάτωση των Ρωμά σε όλε τι ε, χώρε μέλη και επίση δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διάκριση όπω γίνεται πολύ συχνά. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγεία ε, στη συνεχή εκπαίδευση και στην επαγγελματική ανακύκλωση είναι ικανέ και αναγκαίε συνθήκε προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση σε αξιοπρεπή εργασία. Και η συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών είναι επίση απαραίτητη γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να συμμετέχουν και οι τοπικές αρχές. Ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί σα μιλώ. Τα πάντα για αυτού, αλλά τίποτα χωρίς αυτού. Και εδώ ε, στο Κοινοβούλιο υπάρχουν εξαιρετικοί ε, Ρωμά Ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ κύριε Διασδεμέρα. Για 1,5 λεπτό η κυρία Γκόγκ. Ευχαριστώ πρόεδρε η δεύτερη σύνοδο κορυφή στην Κόρδοβα δίνει μια, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να καταμετρήσουμε τι εξελίξει που είχαμε την τελευταία τριετία και να τι αξιολογήσουμε να δούμε πώ βελτιώθηκαν οι ζωέ, καθώ και η κοινωνική ένταξη, αυτή τη πλέον ευάλωτη εθνοτική μειονότητα, στον Ρωμά, τη πλέον ευάλωτη σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να γίνει ένα, αυτό το θέμα ένα θέμα ευρωπαϊκών διαστάσεων και όχι μόνο να απασχολεί τα κεντρικά θεσμικά όργανα τη Ευρώπη. Χρειαζόμαστε εδώ συνολικέ λύσει. Πρέπει να λάβουμε τα απαραίτητα βήματα και από τις πλευράς του Κοινοβουλίου έχοντας εγκρίνει το ψήφισμα να προτείνουμε μάλλον το ψήφισμα που ακόμη δεν έχει ε, εγκριθεί και να λάβουμε περισσότερα βήματα. Βήματα κατά τη θητεία της ε, Ενεργεία Επιτροπής. Στην τελευταία μας έκθαση για την αγορά εργασίας και την κοινωνική κατάσταση το Ρωμά ε, είδαμε ότι έγιναν εκεί πολύ σημαντικέ διαπιστώσεις ότι η καταπολέμηση της ένδυα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να συνδυαστεί με όλη αυτή την προσπάθεια. Και τώρα θα πρέπει να δούμε πώς τα ευρωπαϊκά κονδύλια κατά διάφορα ταμεία συνέβαλαν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρωμά πώς βελτιώσαμε την, ε, πώς διευκολύναμε την κοινωνική τους ένταξη. Εδώ απαιτούμε πληροφορίες και στοιχεία. Γνωρίζουμε όμως όλοι ότι τα δεδομένα για τις εθνοτικές μειονότητες είναι πάντοτε ευαίσθητα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον χειρισμό και την διαχείριση των δεδομένων αυτών. Τώρα για τις διάφορες δράσεις και ενέργειές μας θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπήρξαν προβλήματα το Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό. Το λόγο έχει η κυρία Κιλ Νίλσεν. Το ζήτημα το Ρωμά είναι πολύ έντονο στην περιφέρειά μου, στη Δυτική Γαλλία. Στην Άντι πάνω από χίλιοι ε, διώκονται γιατί δεν έχουν που να τους δεχθούν. Τους στέλνουν από τη μια στην άλλη περιφέρεια, στην Έντρα, στη Ροζέ, ε, στην ευρύτερη ε, περιφέρεια της Νάντης. Οι άνθρωποι αυτοί περιπλανώνται γιατί δεν μπορεί κανείς να τους εξασφαλίσει διαμονή. Οι απαντήσει δεν μπορούν να είναι τοπικέ, πρέπει να είναι συνολικέ Να συμπεριλάβουμε αυτή την πολιτική σε όλε τι πολιτικέ τη Ένωση για να μην υφίστανται αυτοί οι Ευρωπαίοι πολίτε τέτοιε διακρίσει. Από την άλλη θα ήθελα να σε ψήσω την προσοχή στην ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών. Το πρόβλημα των γυναικών Ρωμά είναι τεράστιο. Ε, βία ενδοοικογενειακή, ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, ε, μία στις δύο γυναίκες, 43% στα 22, έχει ήδη υποστεί έκτρωση σύμφωνα με ε, τους ε, γιατρούς χωρίς σύνορα. 17 ετών αποκτούν το πρώτο τους παιδί. Πολύ λίγες έχουν ε, πρόσβαση και καταφεύγουν στην αντισύλληψη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το ζήτημα των γυναικών και προτεραιότητα η παιδεία θα πρέπει να τους ευαισθητοποιήσουμε για τα θεμελιώδη τους δικαιώματα, να τους ευκολύνουμε την πρόσβαση στις κοινοφελείς υπηρεσίες και ελπίζω η δεύτερη αυτή σύνοδος κορυφής να αποδείξει τη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει αυτό το θέμα συνολικό και παγκόσμιο. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό κύριος Φοντάνα. Grazie, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα των αρωμά γίνεται ένα και πιο πολύπλοκο και χρειαζόμαστε αποτελεσματικές λύσεις. Οι εκπρόσωποι τους, τα θεσμικά όργανα, η κοινωνία των πολιτών ζητούν να συμπεριληφθούν στον κοινωνικο-οικονομικό ιστό. Ο Σπανίος όμως αναφέρεται το βασικό σημείο, δηλαδή ότι η ένταξη είναι μια ιστορική και πολιτισμική διαδικασία διμερούς χαρακτήρα. Χωρίς να υπάρχει διάθεση από πλευράς των Ρωμά να δεχτούν τους κανόνες και τον πολιτισμό των χωρών στις οποίες διαμένουν και χωρίς να απαρνηθούν όλες αυτές τις συμπεριφορές οι οποίες δεν συνάδουν με την ε, ε, ειρηνική συνύπαρξη, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ενσωμάτωσή του. Όσο και να αναθέτουμε κονδύλια και να γίνεται χρηματοδότηση, δεν θα έχουμε ουσιαστικές λύσεις. Η πρόκληση δεν αντιμετωπίζεται με δημαγωγίες. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα με ρεαλισμό και να συνειδητοποιήσουμε ότι η συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία και τα θέματα των θέσεων απασχόλησης θα αποτελέσει βασικό στοιχείο στην ένταξη των Ρωμά στην αγορά εργασίας. Όπως μας διδάσκει η ιστορία, η δύσκολη ενσωμάτωση δεν θα μπορεί να είναι... Ε, μόνο λόγω των χωρών υποδοχής. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, ευθύνε και προς τις δύο πλευρές. Ευχαριστώ πολύ. Για δύο λεπτά ο κύριος Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω την ε, να στηρίξω εδώ την συγκεντριά μας που εργάστηκε τόσο σκληρά για το θέμα αυτό και για την κατάσταση των ε, πληθυσμών ε, Ρώμα στην, Ρωμά στην Ευρώπη. Εδώ δεν αφορά το θέμα αυτό μια επιμέρους ευρωπαϊκή χώρα, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωμά είναι μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν και εμεί να αξιολογήσουμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούμε πώ μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάστασή του. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση άκουσα την Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγεί ποιες είναι οι θέσεις της Επιτροπής. Νομίζω ότι τη στιγμή αυτή είναι η καταλληλότερη δεδομένης και της ε, Συνόδου Κορυφής που θα οργανωθεί στην Κόρδοβα τον ερχόμενο μήνα. Η κατάσταση δεν μπορεί να παραμείνει ως έχει, διότι δεν πρόκειται να λυθεί από, μόνο του το πρόβλημα. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι καλού μπορούμε για να βγουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι πληθυσμοί από το περιθώριο και από την ε, συνθήκε ε, ένδυας τις οποίες ζουν. Κατά συνέπεια θα πρέπει να λάβουμε τέτοια μέτρα ώστε να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ευκαιρίες που ισχύουν και για τους υπόλοιπου Ευρωπαίους πολίτες. Ιδίω να ξεφύγουν από την ανεργία, να μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, η ζωή τους να γίνει πλέον αξιοπρεπής και να τους δοθούν ευκαιρίες εργασία. Χωρίς αυτά δεν μπορούν να προχωρήσουν, αλλά με τέτοια μέσα και θα μπορέσουν να στηρίξουν τους εαυτούς τους και να συντηρηθούν, αλλά και να ωφελήσουν γενικότερα την κοινωνία. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε τα απαραίτητα βήματα για να έρθουν οι φραγμοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τους πληθυσμούς Ρωμά. Και ελπίζω ότι το μήνυμα που θα στείλει το Ευρωκοινοβούλιο μας θα είναι ένα μήνυμα αλληλεγγύης προς τους, προς τους Ρωμά. Ένα μήνυμα που θα υιοθετηθεί και στην επόμενη Συνοδό Κορυφής. Ευχαριστώ κύριε Μπουσουτήλ. Το λόγο τώρα έχει για 1,5 λεπτό η κυρία μου η Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δέκα εκατομμύρια ε, Ρωμά τσιγκάνοι ζουν στην Ευρώπη. Ε, ε, αντιπροσωπούσαν αν ήταν κράτος ένα κράτος μεσαίου μεγέθους. Δεν είναι όμως κράτος. Ο, Γκανικό λαό πάντα έβαζε πάνω από κάθε σύνορο την ευρωπαϊκή του διάσταση. Γι' αυτό είναι και πολίτε δευτέρα κατηγορία και υφίστανται διακρίσει όχι μόνο στην παιδεία, στην υγεία ή στη στέγη, αλλά και ως μετακινούμενοι ε, ε, πληθυσμοί που είναι η ίδια τους υπεμπτουσία το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει μια, μια Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που λέει ότι οι μετανάστες τσιγκάνοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υφίστανται την ίδια μεταχείριση με άλλους Ευρωπαίους μετανάστες και αυτό είναι κατάφορη παραβίαση ε, του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας. Εμείς οι σοσιαλιστές θέλουμε μια Ευρώπη όπου να γίνονται δεκτές, να αναγνωρίζονται και σεβαστές οι ε, μειονότητες και οι εθνικές σε μια ε, Ευρώπη ελευθερίας δικαιοσύνης και χαιρόμαστε για την οδηγία μη διάκρισης παντού. Σε μια οδηγία που δεν υποστήριζαν εδώ μέσα πάντα όλες οι πολιτικές ομάδες και καλωσορίζουμε και το πρόγραμμα της Ισπανικής Προεδρίας γιατί το θεωρούμε σημαντικό. Δεν ε, επιτρέπονται επιπλέον καθυστερήσεις και ολιγορίες ε, για την ε, υποστήριξη των Ρωμά. Ε, είναι μεγάλη ευκαιρία λοιπόν η Ισπανική Προεδρία και η Σύνοδος Κορυφής της Κόρδοβα για τους Ρωμά ε, και να σπάσει ο ρατσισμός και η σιωπή των ετών αυτών. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει για ένα λεπτό ο κύριος Ρωμέβα. Thank you, Mr. President. There is very little... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ λίγα μπορώ να προσθέσω. Απλώ θα ήθελα να ζητήσω κάτι. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι η Σύνοδο Κορυφή των Ρωμά ήταν πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου μα και κατατέθηκε κατά τη διάρκεια της Σλοβενικής Προεδρίας με στόχο να ε, συγκεντρωθούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και να συζητήσουν για τα θέματα των Ρωμά. Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν για να είναι πιο δραστήριο το κοινοβούλιο μας. Αν όλα τα κράτη-μέλη δεν παραδεχθούν ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση των Ρωμά, ε, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε λύσεις. Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την ένταξη των Ρωμά Τη χρειαζόμαστε αυτή τη στρατηγική, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει την αξιοπιστία της σε διεθνές επίπεδο. Πολλές ε, χώρες ε, δείχνουν το δάκτυλο προ εμάς, διότι ακριβώς ε, δεν αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό. Πρόκειται για ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικής ένταξη και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι και θέμα πολιτική. Είναι πολιτική η συζήτηση και θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση μια για πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ρωμάδα Γουέδα. Για δύο λεπτά η κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ. Η ε, μειονότητα το Ρωμά είναι από τις μεγαλύτερες αλλά και τις πιο ευάλωτες μειονότητες στην Ευρώπη. Γι' αυτό ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα προβλήματά τους. Τη διάκριση, τη φτώχεια, τη μικρή πρόσβαση στην παιδεία, τον αποκλεισμό, την ανεργία. Είναι τεράστια προβλήματα και πολύ συχνά ε, για τους Ρωμά. Δεν θα πρέπει όλα αυτά να οδηγήσουν στον κοινωνικό τους αποκλεισμό. Χρειάζεται ένα ενσωματωμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που να ε, στον πολιτισμό και στις αξίες των Ρωμά. Επιπλέον, να λαμβάνεται υπόψη ελεύθερη κυκλοφορία Τα παιδιά ε, είναι το 46% του πληθυσμού. Γιατί υπάρχει υψηλός δείχτης γεννήσεων και ε, δυστυχώς και ε, η... το προσδόκιμο ζωής τους είναι χαμηλό. Γι' αυτό είναι τόσο πολλά τα παιδιά. Η πρόσβαση παντού στην κοινωνία είναι πολύ σημαντικό και για τα παιδιά. Πολλέ φορές τα παιδιά τους δεν πηγαίνουν σχολείο ή πηγαίνουν, το εγκαταλείπουν πολύ νωρί. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται αυτό το, τη σχολική χρονιά το 2009-2010 ε, το Υπουργείο Παιδείας της ε, Ρουμανίας ε, αποφάσισε να δοθούν 7.483 θέσεις. Ε, ε, γράφτηκαν 2.460 παιδιά και έγιναν δεκτά 2.246. Χρειάζεται προσπάθεια κατέρωθεν και οι ίδιοι θα πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους. Η έλλειψη μόρφωσης τους εμποδίζει να συμμετέχουν με ενεργό τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και ε, πολιτική ζωή της χώρας. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τους βοηθήσει μέσω διαφόρων προγραμμάτων χρηματοδότηση όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Πρόγδες και Νεολαία σε Δράση. Ευχαριστώ κυρία Μπασέσκου. Για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Μποσκούρτ. Thank you, Chair. Roma... Ευχαριστώ. Η Ρωμά, η μεγαλύτερη μειονότητα στην Ευρώπη, ε, υποφέρουν από ρατσισμό, αντιτσιγκανισμό, κοινωνικό αποκλεισμό, ε, διαχωρισμό στα συστήματα της στέγης, της κοινωνικής ασφάλισης κτλ. Οι βραχυπρόθεσμες λύσεις δεν απαντούν στο πρόβλημα. Είναι τεράστια και πολύ διαδεδομένα τα προβλήματα. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε τις υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές, καλές πρακτικές, καθώς επίσης και τα αρνητικά των διακριτικών μεταχειρήσεων. Ένα παράδειγμα, ε, όχι το μοναδικό είναι ότι ε, τους διαχωρίζουν από τις οικογένειές τους και τους βάζουν σε ξεχωριστά ιδιωτικά σχολεία. Μα αυτό είναι επιπλέον διαχωρισμός και επιπλέον ε, ε, ανητική επιρροή στις ζωές των οικογενικών αυτό. Χρειάζεται μια στρατηγική μακροπρόθεσμη, συνεκτική, συλλογική, καλή ευκαιρία της Κόρδοβα είναι διαφορετική από την πρώτη ε, σύνοδο γιατί δεν είχαμε ε, πολιτική δέσμευση ουσιαστική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, καλά θα έκανε να δίνει περισσότερες θέσεις στους Ρωμά αξιώματα και να τους συμπεριλαμβάνει στην κοινωνία. Ευχαριστώ για δύο λεπτά η κυρία Χιούμπνα. Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι, η Σύνοδος Κορυφής της Κόρδοβα θα είναι μια δοκιμασία για όλους εμάς, για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και για τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να δείξει με σαφήνεια τις ευρωπαϊκές θεσμεύσεις για να δούμε κατά πόσον μπορούμε να έχουμε μια ε, πλήρη και συνολική στρατηγική και να ξεπεράσουμε ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν απλώς με τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά να έχουμε πραγματική οικονομική και κοινωνική ένταξη των Ρώμα. Χρειάζεται εδώ μια κοινή στρατηγική, μια νέα στρατηγική ένα πρόγραμμα δράση για όλα τα σχετικά ζητήματα, τα οικονομικά, τα κοινωνικά και ούτω καθεξής. Πολλά έχουν γίνει και πολλά είναι τα επιτεύγματά μα. Όμω ακόμη ο δρόμο είναι μακρύ. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη, το Κοινοβούλιο, αλλά όπω είπε και ο κ. Λόπε Γκαρίντο και οι περιφερειακέ και τοπικέ αρχέ πρέπει να συνεργαστούν χέρι με χέρι να προχωρήσουν σε αυτό το μακρύ δρόμο. Και είναι, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει συγκεκριμένε ευθύνε για τα θέματα αυτά, να υπάρξει συγκεκριμένη η μορφή συνεργασίας μεταξύ των ε, υπηρεσιών. Το πρόγραμμα δράσης 7 εκατομμυρίων ε, που υλοποιείται αυτή τη στιγμή από την Επιτροπή θα προσπαθήσει να φέρει περαιτέρω αποτελεσματικές λύσεις στα πιο επίγοντα ζητήματα, την εκπαίδευση των νέων παιδιών, την οικονομική ένταξη και να επιτρέψει να, να έχουμε πρόοδο στα ζητήματα τη κοινωνική εκπαίδευση και τη αξιολόγηση. Εδώ η περιφερειακή πολιτική θα πρέπει να μα ενισχύσει και η Επιτροπή να βελτιώσει την τοπική και περιφερειακή συμμετοχή για να διευκολυνθεί ακριβώ η οικονομική και κοινωνική ένταξη των πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων των Ρωμά. Η πολιτικοί μα, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν δείξει τη δέσμευσή του για τα θέματα αυτά. Αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε τι προσπάθειές μα. Η ένταξη των Ρωμά θα είναι κάτι που θα πρέπει να το προωθήσουμε περαιτέρω να γίνει η ευρωπαϊκή αγορά πραγματικά μια αγορά ισότιμη για όλους τους πολίτες. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις απειλές που έχει η δημογραφία και το δημογραφικό ζήτημα για την Ευρώπη. Εδώ λοιπόν πραγματικά υπάρχουν σοβαρού, σοβαροί λόγοι και κίνητρα για την πραγματική κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Ταμπάτσι. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη πραγματοποιήσει μια πρώτη σύνοδο ε, για το θέμα αυτό. Εγώ υπήρξα εισηγητή τότε για το ζήτημα και πρέπει να πω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο πολύπλοκα ζητήματα για την Ευρώπη. Δεν ζηλεύω την Επίτροπο εδώ για την θέση στην οποία βρέθηκε. Πραγματικά αυτό το θέμα είναι περίπλοκο και αφορά όλου μα. Η Ρωμά δεν είναι απλώ μια εθνική μειονότητα, ούτε μια εθνική μειονότητα. Δεν περιορίζονται στα σύνορα ενό κράτου μέλου. Μιλάμε για μια διαφορετική κοινωνική πραγματικότητα. Ωστόσο, οι κοινωνικέ ευθύνε είναι ε, κάτι που δεν έχει. Ε, διανεμηθεί κατά τρόπο ισότιμο μεταξύ των ε, μελών της κοινότητας και των διαφόρων κρατών μελών. Οι κοινωνικές μειονότητες όμως έχουν και αυτές τις ευθύνες τους. Και οι Ρωμά θα πρέπει να ε, ενταχθούν χωρίς όμως να ε, μην αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους. Εδώ δεν μιλάμε για ένα ζήτημα απλώς δημοσιονομικό ή ζήτημα χρηματοδοτικό. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, με πρόσωπα τα οποία πρέπει να ενταχθούν στην κοινωνία της πλειοψηφίας. Και αυτή είναι η Ρωμά. Ω υπήκο ε, κράτου, μέλο που έχει μεγάλη, μεγάλο πληθυσμό Ρωμά στην επικράτειά του, πρέπει να πω ότι πρέπει όλοι οι πολιτικοί άντρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με κυβερνητικέ οργανώσει και οι τοπικοί πολιτικοί να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια. Φυσικά χρειάζονται εδώ κονδύλια, αλλά τα πάντα θα εξαρτηθούν από τη δράση των τοπικών κοινοτήτων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για δύο λεπτά η κυρία Αντωνέσκου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η οικονομική και η κοινωνική ανάπτυξη των Ρωμά αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης. Δεν ξέρουμε ακριβώ ποιο είναι ο αριθμό των Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμω που γνωρίζουμε είναι ότι είναι η φτωχότερη ε, διαμεθοριακή μειονότητα δεν αρκούν οι εθνικές πολιτικές για να αλλάξει η κατάσταση των Ρωμά. Θα πρέπει να αναλυφθούν ευθύνε ε, για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης ε, από κάθε κράτος μέλος, αλλά θα πρέπει να γίνει με συνολικό και συντονισμένο τρόπο οι νέε γενναίε είναι κατ' εμέ ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζουμε. Πρόκειται για ένα πληθυσμό ο οποίο αριθμεί πολλούς νέους ανθρώπους ε, κάτω των 20 ετών στην πλειονότητά του και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει πολιτικές ε, διότι αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα οι διαφορέ μεταξύ των ε, νέων Ρωμά και των υπολείπων πληθυσμών θα αμβληθούν. Ε, θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένε πολιτικές και η πλειονότητα των νέων και των παιδιών ε, Ρωμά θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτές τις αλλαγές. Η βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να ξεκινήσει από μια γενεά παιδιών που θα έχουν πρόσβαση σε παιδεία και υγεία και θα πρέπει ε, να την χάνουν τη ίδια μεταχείρισης με, με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένοι στόχο. Σας θα μπορούσατε να μιλήσετε λίγο πιο αργά, λέει ο πρόεδρο. Θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένε αλλαγέ διότι αλλιώ εκατομμύρια νέων Ρωμά θα είναι περιθωριοποιημένα για όλη του τη ζωή. Η μόνη ελπίδα λοιπόν είναι η κοινότητα αυτή να μην βρίσκεται σε μια ε, κατάσταση ανασφάλειας, διότι θα πρέπει να τους δοθεί μια πραγματική δυνατότητα να αλλάξουν τις ευκαιρίες που τους δίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη και την αλληλεγγύη. Θα πρέπει να εφαρμοστούν συγκεκριμένα ευρωπαϊκά μέτρα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστούμε κυρία για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, συνάδελφοι, Βάσει μιας πρόσφατης δημοσκόπησης, το 76% των ε, Τσέχων υπηκών δεν θέλουν να έχουν ε, γείτονες Ρωμά. Τα τελευταία χρόνια του πολιτικού μου βίου που συμμετείχα σε ένα δημοτικό συμβούλιο της χώρας μου ασχολήθηκα ακριβώς με ζητήματα που είχαν να κάνουν με τις σχέσεις μεταξύ Ρωμά και ε, των υπόλοιπων μελών της κοινωνίας, μη Ρωμά, κατοίκων δηλαδή. Το πρόβλημα δεν είναι τα κονδύλια, δεν είναι το χρήμα. Δεν μπορούμε μόνο με αυτά να βελτιώσουμε την κατάσταση των Ρωμά. Το μόνο που μπορεί να βοηθήσει πραγματικά τα πράγματα να αλλάξουν μακροπρόθεσμα είναι οι Ρωμά να ενταχθούν στην κοινωνία ως ισότιμοι πολίτες, σε μια ευρύτερη κοινότητα. Όμως αυτό είναι μια αμφίδρομη διαδικασία. Θα πρέπει οι Ρωμά να αισθάνονται ότι ανήκουν και αυτοί στην κοινότητα στην οποία εντάσσονται και να ε, υποβληθούν βεβαίω και να σεβαστούν τα ισχύοντα τοπικά πρότυπα. Ο πληθυσμό που αποτελεί την πλειοψηφία θα πρέπει επίση να δίνει ένα παράδειγμα στου Ρωμά. Πρέπει να έχουμε μία, έναν ε, συνολικό αγώνα, έναν ε, επίμονο αγώνα κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Τέτοια φαινόμενα είναι απαράδεκτα και αυτό να αποτελέσει τη βάση μας για το μέλλον. Ευχαριστούμε. Η κυρία Σάμπου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από την αρχή θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα μου. Ελπίζω να επιτύχει η ε, Σύνοδος Κορυφής της Κόρδοβας για να υπάρχει μια κοινή στρατηγική για επίλυση ε, των προβλημάτων της κοινότητας των Ρωμά. Είναι μεγάλες οι διακρίσεις. Παρά τα χρήματα που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια για τη βελτίωση της κατάστασής τους, και πρόκειται για πολλά ε, χρήματα, 500 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, καλό είναι να περάσουμε από τις καλές προθέσεις στις καλές πράξεις. Ε, δυστυχώς όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα δεν έχει επιδείξει την απαραίτητη πολιτική βούληση για συντονισμό ε, της πολιτικής για συμπερίληψη των Ρωμά στην κοινωνία και καταπολέμηση των ρατσιστικών επιθέσεων που δέχονται και διακρίσεων. Θα πρέπει αυτό το θέμα να το δούμε ξεχωριστά ε, και συγκεκριμένα ο Επίτροπος Κοινωνικών Υποθέσεων να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Να εργαστεί προς την κατεύθυνση αυτή με συμμετοχή ειδικών ε, που να προέρχονται από την εθνότητα το Ρωμά. Χρειάζεται ε, πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μην δεονίζονται οι ε, ανισότητες που έχουμε και στον αναλφαβητισμό και ε, στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό ζητώ από την Εκτελεστική Επιτροπή να ψυχώσει ε, και προγράμματα συμμετοχή στην αγορά εργασία στον Ρωμά, σε συνεργασία με τι ίδιε κοινότητε του, τι τοπικέ κοινωνίε, για να υπάρχει και καλύτερη συνεννόηση και συντονισμό και συνεργασία με τι ΜΚΟ. Ευχαριστώ. Διαδικασία Catch the Eye. Και θα είμαι πάρα πολύ αυστηρό με το χρόνο διότι ε, έχουμε καθυστέρηση. Ο κύριος Πέρ για ένα λεπτό πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, το γεγονός, μάλλον θα ήθελα σίγουρα να σας συγχαρώ που προβλέψατε αυτό το σημείο για συζήτηση, την Σύνοδο Κορυφής δηλαδή για τους Ρωμά, τη δεύτερη Σύνοδο Κορυφής, διότι ακριβώς αυτό δείχνει τη σημασία που προσδίδουμε στο όλο θέμα. Επίσης αποδεικνύουμε ότι όλες οι πολιτικές ομάδες και παρατάξεις έχουν ενεργό συμμετοχή στην εξέταση του θέματος μας απασχολεί όλους και βεβαίως θα προετοιμαστούμε έτσι καλύτερα για να έχουμε μια ισχυρότερη στρατηγική προκειμένου να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα το Ρωμά. Εδώ ε, φυσικά πρέπει να δούμε και τι νομικά μέτρα μπορούμε να λάβουμε, γιατί σίγουρα υπάρχει και η αρμοδιότητα των επιμέρους κατομελών, όμως θα χρειαστεί να ανταλλάξουμε πληροφορίες, δεδομένα και καλές πρακτικές. Εγώ έρχομαι από την Σλοβενία, όπου έχουμε ένα ε, Ινστιτούτο για τους Ρωμά, που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των δημόσιων αρχών και των γονιών ή των παιδιών και αυτό βελτιώνει την ένταξη των παιδιών στο σχολείο. Πέντε ομιλητές μόνο, η ε, κυρία Κρέτσου. Ο κύριος Παπα-Νικολάου, ο Γκουρ Μαρινέσκου και άλλοι δεν θα έχουν χρόνο να μιλήσουν. Στη διαδικασία κάτσε. σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Η κυρία Κρέτσου, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η πρώτη σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Ρωμά αναγκάστηκε να αναγνωρίσει την αποτυχία των κρατών μελών ε, για τη εγγύηση των δικαιωμάτων των Ρωμά και κατέδειξε την ανάγκη να υπάρχει μια, μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Δυστυχώς παραμένει τεράστια η ε, διαφορά ανάμεσα στα λόγια και στα έργα. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση των ανθρώπων αυτών που είναι και η μεγαλύτερη πλέον μειονότητα στην Ευρώπη που έχει μεγαλύτερη φτώχεια και το μεγαλύτερο κοινωνικό αποκλεισμό. Οι προοπτικές δυστυχώς δεν είναι πάρα πολύ αισιόδοξε. Η μισή ε, Ρωμά είναι ανήλικη. Γιατί ε, ε, είναι μεγάλος, είπαμε, ο δείκτης γεννήσεων και μικρό το προσδόκιμο ζωής στον Ρωμά. Θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί και τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην παιδεία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να επέλθουν οι αλλαγές που θέλουμε, να μπουν στην αγορά εργασίας και να βγουν από το φαύλο κύκλο της κοινωνικής απομόνωσης και αποκλεισμού. Ευχαριστώ. κύριος Μάκουλα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι Ρωμά εκπροσωπούν μία κοινότητα πολιτιστική και εθνοτική που ξεπερνά τα σύνορα των επιμέρου γύρω στα 10 εκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη και παραπάνω. Πρέπει εδώ λοιπόν η δράση των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι συντονισμένη και συνολική. Ήδη έχουμε λάβει σημαντικέ πρωτοβουλίε ω τώρα για το θέμα αυτό, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε, να έχουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή στρατηγική για του Ρωμά. Δράσει πραγματικά στοχοθετημένε και τακτικέ ε, συστηματικέ μελέτε αντικτύπου. Είναι πολλά τα κράτη που φιλοξενούν πληθυσμού Ρωμά στην επικράτειά του. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό έχει ευρωπαϊκέ διαστάσει. Πριν την ένταξη τη χώρα μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρουμανία είχε προβλέψει μια στρατηγική για τη βελτίωση τη διαβίωση των συνθηκών διαβίωση στο Ρωμά. Για παράδειγμα, προβλέφθηκαν υποτροφίε κάποιε φορέ για φοιτητέ Ρωμά στα κρατικά πανεπιστήμια. Και αυτό βεβαίω βελτίωσε τι δυνατότητε φίτηση των ε, νεαρών της κοινότητας αυτής και τις δυνατότητες και προοπτικές ε, κοινωνικής τους ένταξης, συμπερίληψής τους στην αγορά εργασίας, καταπολέμησης της ένδυας και πρόσβαση ε, πρόσβασης στις υγειονομικές υπηρεσίες. Χρειάζεται όμως εδώ μια συνεκτικότερη και συνολικότερη ευρωπαϊκή στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Η κυρία Μορβάη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε τα τσεγκανόπουλα ή τα παιδάκια των Ρωμά θέλετε έχουν ως μόνο τρόπο να βγουν από την κατάστασή τους το σχολείο, συστηματικά, την παιδεία. Είναι κρίμα που το πολιτικά ορθόν δεν μας επιτρέπει να επεμβαίνουμε. Αφήνουν τους γονείς ε, να μην στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο γιατί πολλές φορές διαφωνούν οι γονείς με το να πάνε τα παιδιά σχολείο. Αυτό είναι πολύ ε, μεγάλη διάκριση ει βάρο των κοριτσιών κυρίω. Γιατί πολλές φορές οι ε, γονείς ε, τους αναθέτουν την ανατροφή των αδελφών τους, τον οικοκυριών, της ζωή του σπιτιού, αντί να τα στέλνουν στο σχολείο. Καλές οι νομικές ε, διατάξεις και οι κανόνες, αλλά θα πρέπει να κάνει κάτι και το κράτος για να προστατεύει τα παιδιά αυτά και να επιβάλλει κυρώσεις, να τιμωρεί τους γονείς αυτούς που δεν αφήνουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν στο σχολείο. Να τους αφαιρούν τα επιδόματα και τα λοιπά. Εκπαίδευση, παιδεία. Ευχαριστώ κυρία ε, Σμόκοβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Είναι η πιο ευάλωτη μειονότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ρωμά. Γι' αυτό θεωρώ ότι όλα ε, τα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε για να τους βοηθήσουν να είναι ευπρόσδεκτα, να συμμετέχουν στην κοινωνία, στην οικονομία. Το κλειδί περνάει μέσα από την εκπαίδευση και τη μόρφωση. Και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να καταργηθεί ε, η διάκριση, κάθε είδους διάκριση, ε, καλυμμένη και ανοιχτή. Επίσης θέλω να συζητάμε ειλικρινά αυτά τα θέματα, να μιλούμε για τα δικαιώματα των παιδιών, των Ρωμά. Τα δικαιώματα αυτά τα παραβιάζουν οι γονεί του οι ίδιοι. τους αρνούνται τη δυνατότητα να ε, ε, προκόψουν στη ζωή τους. Ε, θα πρέπει στην αναζήτηση τη λύση να συμμετέχουν και ήδη οι Ρωμά για τη μόρφωση, για την εκπαίδευση των παιδιών, για την ανατροφή των παιδιών, για τη βελτίωση την ίδια των ε, ε, συνθήκων διαβίωσης. Εγώ που δεν θέλω να γίνω επίτροπος, δεν έχω τέτοια φιλοδοξία, πρέπει να πω το εξής. μιλάμε για μια σύνοδο κορυφής εδώ, ε, που έχει και κοινωνικά στοιχεία και κοινωνικά επιδόματα. Να τα συζητήσουμε και αυτά. Ευχαριστώ. Ε, ζητώ συγγνώμη για εκείνους που ζήτησαν το λόγο για το ΚΑΤΣΙΑΕ, αλλά έχουμε ένα τέταρτο ήδη καθυστέρηση για τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή. Ο κύριος Λόπες Γαρίδο, εξ του Συμβουλίου. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση που έγινε για την κοινότητα των Αθήγκανων, για την Σύνοδο Κορυφής ε, της Κόρδοβας, καταδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η κοινωνική ένταξη και η οικονομική ένταξη των Αθήγκανων είναι ένα πρόβλημα με τεράστιες διαστάσεις που απαιτεί και ευρωπαϊκή στρατηγική. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε μετά από κάποιες προόδους οι οποίες έγιναν αλλά δεν αρκούσαν ε, στη διάσκεψη της Κόρδοβας η οποία ακούστηκε πολλές φορές σήμερα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο εργασίας ε, το οποίο θα τηρήσει το Συμβούλιο και θα πρέπει το ε, σχέδιο εργασίας αυτό να εκπονηθεί στα πλαίσια του προγράμματος της Τρόικας να είναι ένα πρόγραμμα δράσης, ένα πρόγραμμα εργασίας το οποίο θα θεωρεί ως ένα από τα πιο σημαντικούς του πυλώνες ε, τα διαρθρωτικά ταμεία και να έχουμε κοινωνική συνοχή και ένταξη καθώς ταυτόχρονα να συγκεκριμενοποιηθεί και σε συγκεκριμένες δράσεις. Δράσεις οι οποίες κατά την άποψή μου θα πρέπει να είναι αφενός ε, δράσεις που θα στοχεύουν σε συγκεκριμένα προβλήματα της κοινότητας των Ρωμά, τις διακρίσεις, ε, που αντιμετωπίζει παραδείγματο χάρη πρόβλημα σε πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες ή στην παιδεία, προβλήματα των γυναικών που πλήττονται από την ένδυα, ε, δεν υπάρχει στέγαση επαρκής, ε, προβλήματα διάκρισης ή βία Στην περίπτωση των νέων αυτή τη στιγμή με την οικονομική κρίση, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένε δεξιότητες για τους νέους Ρωμά και δυσχεραίνει η πρόσβαση σε θέσεις εργασίας ή τα παιδιά τα οποία όπως ακούσαμε έχουν ένα προσδόκιμο ζωής 10 ε, χρόνια μικρότερο από αυτό που έχουν ε, τα παιδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά μέσο όρο. Και επίσης θα πρέπει να έχουμε και κάποιες δράσεις οι οποίες θα ευνοήσουν την ίδια την κοινότητα των Ρωμά. Επειδή είναι μία από τις κοινότητε η οποία αντιμετωπίζει τις περισσότερες διακρίσεις, οτιδήποτε κάνουμε κατά των διακρίσεων θα είναι υπέρ του. Όσον αφορά τώρα στι γενικευμένε δράσεις, θα πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν ε, συντομότερο την οδηγία η οποία θα ευνοήσει τις γυναίκες ε, Ρωμά και την οδηγία κατά των διακρίσεων που θα ευνοήσει την κοινωνία των Ρωμά. Και όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω εδώ, θα πρέπει να προσανατολίζονται κυρίως με παταναλιστικό τρόπο διότι θα πρέπει να σεβαστούμε και την ταυτότητά τους και τα συγκεκριμένα πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Κοινοβούλιο για τις πολλές προτάσεις και υποδείξεις που έκανα, Θα ληφθούν υπόψη από τον ε, ε, ε, Επίτροπο Αρμόδιο και εμένα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να δεχτεί σε καμία περίπτωση τη διάκριση και τον αποκλεισμό των Ρωμά από την κοινωνία μας λόγω της ε, εθνικής της προέλευσης. Έχουμε και εργαλεία και πολιτικές. Το θέμα είναι πώς ε, τα εφαρμόζουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε, πώς ε, βάζουμε αυτά τα θέματα στις πολιτικές μας, στα εργαλεία και τα μέσα που έχουμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ούτε ταμείο για τους Ρωμά, ούτε οδηγία για τους Ρωμά. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να λάβουμε υπόψη μας πλήρως τα προβλήματά τους όταν εφαρμόζουμε το κοινοτικό δίκαιο και όταν ε, χρησιμοποιούμε τα κοινοτικά κονδύλια. Συνεργασία, εταιρική σχέση, το είπατε κι εσείς, όλων των πρωταγωνιστών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει την προσέγγιση της στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τη Συμπερίληψη των Ρωμά και ε, στις άλλες ε, εσωτερικές διαδικασίες. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω και κάτι άλλο, σαφέστατα. Βεβαίως ο αποκλεισμό των Ρωμά έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά έχει να κάνει κυρίως με κοινωνικές ψυχές και οικονομικές. Παράδειγμα, θα ήθελα να παραθέσω μια μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας για το οικονομικό κόστος του αποκλεισμού των Ρωμά για να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά τα στοιχεία αυτά. Χρειαζόμαστε να βρούμε λύσεις ε, και αυτό είναι προς όφελος των κοινωνιών μας γενικά. Έτσι λοιπόν, εφαρμογή των μέσων που έχουμε, που διαθέτουμε ήδη με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Για να γίνει αυτό χρειάζεται στρατηγική προσέγγιση, συμπερίληψη ε, αυτών των στοιχείων στις εγκάρσεις πολιτικές, το mainstreaming, συνεργασία, κινητοποίηση των απορριτήτων ε, οικονομικών πόρων και μια στρατηγική να ε, μαθαίνουμε και από τις επιτυχίες και από τις αποτυχίες μας. Αυτό που θα πρέπει να αποφύγουμε είναι να δημιουργηθεί μια στρατηγική στα χαρτιά και μόνο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι αποτελέσματα, συμπερίληψή του στην κοινωνία, στα σχολεία. Πολύ μιλήσατε για τα σχολεία και την μόρφωση. Το σημείωσα. Θα μελετήσω τις λεπτομέρειες ε, της δράσης μας για την προσχολική ηλικία, θα ε, δούμε τι κάνουμε εκεί και στη συνέχεια στην αγορά εργασίας. Εδώ είναι αρμόδιος ο συνάδελφος Άντρο και ε, θα ε, φροντίσει να εντοπίσει ειδικού στόχους και συμμετοχή στην κοινωνία, όπου βεβαίως αυτό είναι θέμα όλων των πολιτικών μας. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει στην επόμενη ε, σύνοδο. Ερχόμαστε τώρα σε ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ορίστε κύριε Ταμπάιτζη. Ευχαριστώ. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα, λέει ο κύριος Ταμπάιτζη. Μόλις διαπίστωσα ότι κλωνοποιήθηκα από το υπολογιστή. Κάποιος άλλος συνάδελφος είχε βάλει την κάρτα του ε, δίπλα στην κυρία Γκέρνς ε, στο έδρανο που δεν είναι δικό μου και γράφει παντού τα Και η συνάδελφος Γκέρνς ε, λέγεται τα ε, κάτι πρέπει να κάνετε γιατί γέμισε το κοινοβούλιο κλόνους του Ταμπάιτζη και δεν αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα. Στείλτε κανένα τεχνικό σας παρακαλώ. Μάλιστα, το σημειώνουμε. Ε, και προχωρούμε στις ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πιο σύντομη σήμερα η συζήτηση αυτή γιατί 25 λεπτά καθυστερήσαμε για λόγους διαδικαστικού. Ζητώ συγγνώμη. Θα τελειώσουμε γύρω στι